πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Η πρώτη είναι η εξής. Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε, επαναλαμβάνω. Η πρώτη ανακοίνωση είναι η εξής. Ο πρόεδρος έχει λάβει από την ομάδα συντηρητικών και μεταρρυθμιστών έτοιμα αλλαγής ε, ονόματος σε επιτροπή και σε αντιπροσωπεία. Οι αλλαγές θα υπάρχουν στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης και αν δεν έχετε παρατηρήσεις να υποβάλλετε πριν την έγκριση των πρακτικών